Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, έχω την ιδιαίτερη χαρά σήμερα να υποδέχομαι τον πρόεδρο του Ισραήλ, κύριο Σιμών Πέρες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μεγάλη τιμή για μας, κύριε πρόεδρε, η επίσκεψή σας σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας και τις ελπίδες σας για το μέλλον. Μεταξύ Ευρωπαίων και Ισραηλινών πολιτών σήμερα υπάρχει πολύ στενός δεσμός και θέλουμε να τον επιβεβαιώσουμε και να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με το μέλλον και με τη σημερινή σας επίσκεψη. Πολιτισμικές όσο και οικονομικές σχέσεις έχουμε όλο και πιο στενές. Κοινή ιστορία πλούσια αλλά και οδυνηρή που θα μας ενώνει ε, για πάντα στενά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ και οι δύο δημιουργήθηκαν μετά από τον τρόμο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά την εμπειρία του ναδύρ της ανθρώπινης ιστορίας, το ολοκαύτωμα. Στην Ευρώπη, εδώ, πάνω από 60 χρόνια στην Ευρώπη, ε, μάλλον πριν από 60 χρόνια στην Ευρώπη, ε, ορκίστηκαν οι πολίτες ε, ποτέ πια. Και αυτό το ποτέ πια σας το λέγει ένας Γερμανός πολίτης που έχει τη μεγάλη τιμή να προεδρεύει σε ένα πολύ εθνικό κοινοβούλιο. Αυτό το ποτέ πια είναι και για μένα και για όλους εδώ νομίζω και σήμερα και για πάντα το ύψιστο καθήκον. Ο αγώνας μας κατά του αντισημιτισμού, του αποκλεισμού, κατά της μη αλλοδοξίας είναι το ίδιο το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είμαστε το Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι το δικαίωμα στην ύπαρξη του Ισραήλ είναι αδιαφυσβήτητο και το δικαίωμα του λαού του ε, να ε, ζει με ειρήνη και ασφάλεια. Είναι αδιαπραγμάτευτα αυτά. Είμαστε βαθύτατα πεπισμένοι ως Ευρωπαίοι και το ξαναλέγω εγώ ως Γερμανός ιδιαίτερα αλλά επιθυμώ, Πρόεδρε, να μπορούσα να πω σήμερα ότι από την περισμένη φορά που συναντηθήκαμε ε, υπάρχουν πρόοδοι ε, στη σύγκρουση ε, της Μέσης Ανατολής. Δυστυχώς μετά από μακρές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις ε, παραμένει ανύπαρκτη μια σοβαρή πρωτοβουλία για την ειρήνη. Ο Παλαιστινιακό έχει, λαός έχει εξίσου δικαίωμα όπω και ο Ισραηλινό, ένα δικαίωμα ε, ανεξαρτησία και ζωή σε ειρήνη και ασφάλεια. Ούτε όμως ο Ισραηλινός ούτε ο Παλαιστινιακός λαός είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια διαρκή ειρήνη. Θέλουμε όλοι να ζήσουμε, να δούμε και τους δύο λαούς να συνεπάρχουν σε δύο δημοκρατικά ε, κράτη με ασφαλή σύνορα και να μπορούν να ζουν σε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας. Το 1993 εσείς Πρόεδρε στο βιβλίο σας για μια νέα Μέση Ανατολή εκφράσατε το όραμά σας ε, για το μέλλον της περιοχής σας. Μια Μέση Ανατολή με οικονομική συνεργασία που να δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων και με τη συμφιλίωση να ε, σφυριλατεί την ειρήνη. Ορισμένοι σας χαρακτήρισαν τότε αφελή. Εδώ στο Κοινοβούλιο εμείς σας χαρακτηρίζουμε θαραλέο, διότι έχετε τα ίδια οράματα και το ίδιο θάρρος που χαρακτήριζε τους ιδρυτές πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοιραζόμαστε μαζί σας το όνειρό σας για τη Μέση Ανατολή, μια ήρεμη και ειρηνική περιοχή και θα σας υποστηρίζουμε και στο μέλλον κύριε Πρόεδρε Πέρες. Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με χαρά θα ακούσουμε την ομιλία σας. Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φίλε μου Μάρτιν Σούλτς, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μεγάλου αυτού σώματος της ελευθερίας και της ειρήνης που έχει μεταμορφώσει την ιστορία της Ευρώπης και το μέλλον όλου του κόσμου μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία και το προνόμιο να μιλήσω ενώπιόν σας. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για όλους μας και για το λαό του Ισραήλ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Στέκομαι μπροστά σας με μνήμες που καίνε την καρδιά μου αλλά και με μεγάλη ελπίδα στην ψυχή μου φέρω τη βαθιά οδύνη του παρελθόντος και βλέπω με εμπιστοσύνη, ατενίζω με εμπιστοσύνη το μέλλον. Ήρθα στο Ισραήλ το 1934 σε ηλικία 11 ετών. Το 1942 οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης όπου γεννήθηκα κάηκαν ζωντανοί. Αν η οικογένειά μου είχε καθυστερήσει για 8 χρόνια τη μετανάστευσή του στο Ισραήλ, θα ήμασταν κι εμείς μεταξύ αυτών που εξολοθρεύτηκαν. Ένα χρόνο πριν από την δημιουργία του Ισραήλ, το 1947, στελεχώθηκα σαν ένας από τους ηγέτες στο αρχηγείο της Χάγκανα. Από τότε το Ισραήλ έτυχε επιθέσεων 7 φορές στα 65 χρόνια της ύπαρξής τους. Ήμασταν λιγότεροι σε αριθμό, λιγότεροι σε όπλα και είχαμε μονάχα μία επιλογή μπροστά μας. Ή να νικήσουμε ή να χαθούμε, να πεθάνουμε. Και εγώ συμμετέσχα στην αντιμετώπιση ενός άλλου εχθρού, της ερήμου. Κερδίσαμε τον αγώνα αυτό κάναμε να ανθίσει η έρημος. Έχω πολλές μνήμες. Έχω όμως και πολλά όνειρα. Δεν ήρθα εδώ για να σας αναφέρω τις αναμνήσεις μου. Ήρθα να συνεχίσω τα όνειρά μου. Οι άνθρωποι οριμάζουν, γίνονται ηλικιωμένοι, αλλά τα όνειρα παραμένουν χωρίς χρόνο. Έχουμε αλλάξει. Η Ευρώπη έχει αλλάξει. Θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μας για τις αλλαγές που γνώρισε η Ευρώπη. Η Ευρώπη μπόρεσε να ξανασταθεί όρθια μετά από δύο από τους χειρότερους παγκόσμιους πολέμους στην ιστορία της. Ξεπέρασε το παρελθόν της, δημιούργησε μια νέα Ευρώπη. Η διχασμένη Ευρώπη των τελευταίων χιλίων ετών μεταμορφώθηκε σε μια ενωμένη σύγχρονη Ευρώπη, τη σημερινή Ευρώπη. Αντιμετωπίσατε το παρελθόν κάνοντας τα στρατόπεδα πανεπιστήμια, χώρους γνώσης. Η Ευρώπη τώρα έχει αναγνωρίσει ότι ο ρατσισμός είναι ένα έγκλημα. Ξέρω ότι αντιμετωπίζετε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Αλλά οι ουρανοί σας δεν έχουν τη σκιά και τα σύννεφα του πολέμου η μια ευρωπαϊκή χώρα ήταν αυτή η οποία εισήγαγε το βραβείο Νόμπελ και τώρα η μια Ενωμένη Ευρώπη δίκαια κατέκτησε το βραβείο Νόμπελ. Η Ευρώπη έχει διορθώσει τα σφάλματά της και οικοδομεί ένα καλύτερο κόσμο. Για μας η Ευρώπη του ολοκαυτώματος του ΣΟΑ γίνεται τώρα η Ευρώπη που υποστηρίζει την αναγέννησή μας. Αγαπητοί φίλοι, η ιδέα της αναγέννησης του Ισραήλ γεννήθηκε στο ευρωπαϊκό έδαφος στα τελευταία χιλιά χρόνια ζούσαν περισσότεροι Εβραίοι στην Ευρώπη από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ήπειρο στον κόσμο. Δυστυχώς δολοφονήθηκαν πιο πολλοί Εβραίοι στην Ευρώπη στα τελευταία 100 χρόνια από ό,τι στις προηγούμενες δύο χιλιετίες. Έχουμε γνωρίσει την χειρότερη τραγωδία της ιστορίας μας εδώ πάλι στην Ευρώπη ονειρευτήκαμε μια αναγέννηση που φαινόταν τότε αδύνατη. Έξι εκατομμύρια Εβραίοι, το ένα τρίτο του εβραϊκού λαού δολοφονήθηκαν στην Ευρώπη. Από την πείνα, από τα, τους θαλάμους αερίου, από τις εκτελέσεις, από τις πυρπολίσεις, μείναν μόνο στάχτες. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι οι δίκαιοι μεταξύ των εθνών ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν μια μικρή αχτίδα φωτός μέσα στο έρευος. Ήταν λίγοι, αλλά ήταν μεγάλοι στον ηρωισμό τους. Το Ισραήλ ξαναγεννήθηκε από αυτές τις τέφρες του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν τότε κάποιος είχε πει ότι μέσα σε τρία χρόνια θα υπήρχε ένα εβραϊκό κράτος, θα τον θεωρούσαν ότι παραλυρεί, ότι είναι ένας παραλυρών οραματιστής και τίποτα άλλο. Τα όνειρά όμως γίνονται πραγματικότητα. Και εξάλλου, αν κάποιος στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε πει την ίδια μέρα ότι μέσα σε έξι σύντομα χρόνια θα μπορούσε να υπάρξει μια νέα ενωμένη Ευρώπη χωρίς σύνορα, χωρίς φραγμούς και πάλι θα θεωρείται ότι είναι στα πλαίσια της μυθοπλασίας αυτό. Και όμως έγινε αυτό το θαύμα. Έξι χώρες υπέγραψαν τη Συνδίκη των Παρισίων και εν καιρό έγιναν μια κοινότητα 27 κρατών από όλη την Ευρώπη. Η σχέση μας λοιπόν και τότε και τώρα είναι ο διάλογος μεταξύ δύο θαυμάτων του ευρωπαϊκού θαύματος και του δικού μας. Το Ισραήλ έχει μία συμφωνία σύνδεσης με την Ευρώπη και έχει στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους σχεδόν τους τομείς. Είμαι εδώ για να σας ευχαριστήσω για τη φιλία σας που βασίζεται σε κοινέ αξίες, στην γεωγραφική εγκύτητα και την κοινή μας ιστορία. Σε πολιτικό επίπεδο, το Ισραήλ είναι μια δυτική δημοκρατία με μεσογειακή εμπειρία θρησκευτικά. Είμαστε το λίκνο των μεγάλων τριών μονοθεϊστικών θρησκειών. Επιστημονικά, το Ισραήλ είναι μια πολύ προχωρημένη χώρα ακόμα και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το Ισραήλ είναι μικρό. Είναι μονάχα το ένα χιλιοστό της επιφάνειας της Μέσης Ανατολής. Είναι το έδαφος μας άγωνο, δεν είναι έφορο, όπως είναι και σε όλη τη Μέση Ανατολή. Λείπει το νερό. Έχουμε μόνο δύο λίμνες, μία είναι η νεκρά θάλασσα και η άλλη και αυτή πεθαίνει. Έχουμε ένα μονάχα ποταμό, τον Ιορδάνη, ο οποίος είναι πλούσιος σε ιστορία, αλλά φτωχός σε νερό. Είμαστε πλούσιοι σε αρχαιολογία, φτωχοί σε φυσικούς πόρους οι μόνοι φυσικοί πόροι που έχουν ανακαλυφθεί από εμά είναι το δυναμικό των ανθρώπων. Είναι ένα παράδειγμα το Ισραήλ μιας χώρας όπου οι πολίτες του έχουν εμπλουτίσει τη γη πολύ περισσότερο από ότι η γη τους έκανε πλούσιους. Ένα παράδειγμα όπου η αφοσίωση των ανθρώπων και η αξία της υψηλής τεχνολογίας έκανε την έρημο να υποταχθεί και να ανθίσει. Περάσαμε 7 πολέμους τους κερδίσαμε όλους. Όταν όμως η ειρήνη έγινε κάτι το εφικτό, ξαναγυρίσαμε όλες τις εκτάσεις και όλα τα στοιχεία που πήραμε από τον πόλεμο στις χώρες οι οποίες έκαναν ειρήνη μαζί μας, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία ειρήνευσης με τους Παλαιστινίους που τους έδωσε τη δυνατότητα και σε μας επίσης να δημιουργήσουμε μια Παλαιστινιακή αρχή. Και μετά αυτό κάτι το οποίο ξεχνούν πολύ, εκενώσαμε τη Λωρίδα της Γάζας. Διαλύσαμε 22 οικισμούς και επαναπατρίσαμε όλους τους επίκους από αυτούς τους οικισμούς. Ήταν μια ευκαιρία για τους Παλαιστινίους να μετατρέψουν τη Λωρίδα της Γάζας σε, ένα ανεξάρτητο, σε μια ανεξάρτητη οντότητα ειρήνης. Αντίθετα και δυστυχώς μετατρέψαν την Λωρίδα της Γάζας σε μια βάση για τρομοκρατία. Δεν ξέρουμε γιατί, δεν ξέρουμε ποιο σκοπό. Ξέρουμε όμως ότι πράγματι αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν επέτρεψε στη διαδικασία ειρήνευσης να προχωρήσει. Το Ισραήλ είναι μια νησίδα σε ένα θυελώδη ωκεανό. Πρέπει να υπερασπιστούμε το νησί μας. Είναι προς το συμφέρον μας να εξασφαλίσουμε ότι θα γαλινέψει η θάλασσα στον περίγυρό μας. Λένε μερικοί ότι αυτό θα χρειαστεί γενιές. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι τέτοιε μεγάλες αλλαγέ μπορούν να γίνουν μόνο σε έξι χρόνια. Ζούμε σε μια νέα εποχή, όταν τα γεγονότα προχωρούν με την ταχύτητα των ε, αεροπλάνων και όχι των αμαξών. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί πολύ σύντομα. Η διαδικασία ειρήνευσης με τους Παλαιστινίους έχει ήδη μια συμπεφωνημένη εκκίνηση και μια τελική λύση η οποία είναι συμπεφωνημένη επίσης. Η λύση είναι δύο κράτη για δύο έθνη. Ένα αραβικό κράτος για την Παλαιστίνη και ένα εβραϊκό κράτος, το Ισραήλ, και τα δύο κράτη να ζουν σε ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική συνεργασία. Τα υπόλοιπα επίμαχα θέματα μπορούν και θα πρέπει να είναι από ε, αντικείμενο διαπραγματεύσεως. Η ειρήνη για το Ισραήλ δεν είναι μονάχα μια στρατηγική επιλογή. Είναι μια κατηγορική επιταγή που προέρχεται από το βάθος της παράδοσής μας. Μετά από την έξοδο, η παράδοσή μας καταδικάζει τη δουλεία και αρνείται την επικυριαρχία γιατί θεωρούμε ότι όλοι είναι γεννημένοι ίσοι. Η παράδοσή μας αυτή λοιπόν μας ζητά να ακολουθήσουμε το δρόμο της ειρήνης. Μαζί με τον εταίρο μου, τον Γίτσα Κράμπιν, που δολοφονήθηκε όπως ξέρετε, εμείς θέσαμε τα θεμέλια της ειρήνης με τους Παλαιστινίους. Και τώρα είναι καιρός να συνεχίσουμε. Να ανανεώσουμε τη διαδικασία ειρήνευσης. Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Παλαιστινιακή Αρχή, να υποστηρίξουμε την οικονομία τους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πλήρη ειρήνη. Υπάρχει μια δύναμη ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής και εσείς και οι Ηνωμένε Πολιτείες την έχουν εκπαιδεύσει και πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους για να αποτρέψουμε την τρομοκρατία και το έγκλημα. Κυρίες και κύριοι, εξακολουθούμε να τίνουμε χείρα ειρήνης προς όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Σε ένα σύντομο διάστημα θα σχηματιστεί μια νέα ελληνική κυβέρνηση. Είναι μια ευκαιρία επανάληψης των διαπραγματεύσεων ειρήνης. Είναι μια ευκαιρία να υλοποιήσουμε τη λύση δύο κρατών. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση ούτε για τους Παλαιστινίους, ούτε και για μας. Δεν είναι μονάχα η δική μας προτίμηση. Είναι αυτό που απαιτεί η τωρινή πραγματικότητα. Η Ορδανία, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις. Απειλούνται και οι τρεις από την τρομοκρατία και χωριστά, μεμονωμένα, αλλά και οι τρεις μαζί οι κοινοί κίνδυνοι πρέπει να οδηγήσουν σε κοινή ασφάλεια. Έχω τη μεγαλύτερη εκτίμηση για τον βασιλιά της Ιορδανίας. Όπως ο πατέρας του έδειξε να είναι θαραλέος και προσιλωμένος στην ιδέα της ειρήνης. Έχω γνωρίζω τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμού Αμπάς για πολλά χρόνια. Και ξέρω ότι καταδικάζει την τρομοκρατία και είναι πραγματικός εταίρος στον αγώνα για την ειρήνη. Και η Ευρώπη εξακολουθεί, όπως υπήρξε στο παρελθόν, να είναι ένας σημαντικός εταίρος για την ειρήνη και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Την επόμενη εβδομάδα θα υποδεχτούμε τον πρόεδρο Ομπάμα στο Ισραήλ ως ένα ιδιαίτερα καλόδεκτο και σημαντικό καλεσμένο. Η υποστήριξή του για την ασφάλειά μας είναι εκπληκτική και η προσήλωσή του στην ειρήνη είναι ακλόντη. Χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε συνεργάζονται για να υποστηρίξουν την ειρήνη και να σταματήσουν να αναχαιτήσουν την τρομοκρατία. Γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ειρήνη στον κόσμο είναι το καθεστώς, το τωρινό καθεστώς του Ιράν. Έγινε μια δικτατορία που είναι δημένη με ένα θρησκευτικό μανδύα. Έχει αναπτύξει μία υπεριαλιστική όρεξη επέκτασης. Κανείς δεν απειλεί το Ιράν. Το Ιράν όμως απειλεί τους άλλους. Θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των αραβικών χωρών. Απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ. Εισάγει λαθρέα όπλα σε πολλές χώρες με στόχο να υπονομεύσει τη σταθερότητά τους. Όχι μονάχα αρνείται το ολοκαύτωμα, αλλά προσκαλεί σε ένα νέο ολοκαύτωμα. Έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν πυρηνικά όπλα και αρνούνται ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους. Μια πυρηνική βόμβα στα χέρια μιας ανεύθυνης εξουσίας όπως αυτή του Ιράν είναι ένας άμεσος κίνδυνος για όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν καταλήξει στα συμπεράσματα αυτά και έχουν οικοδομήσει από κοινού μια πολιτική να αναχαιτήσουν αυτό το κίνδυνο. Γι' αυτό έχετε ορθά <clears throat> αποφασίσει να επιβάλλετε οικονομικές κυρώσεις και έχετε κάνει σαφές ότι εάν το Ιράν δεν απαντήσει σε αυτή την έκκλησή σας, θα υπάρξουν ενδεχομένως και άλλες επιλογές. Εκτός από την πυρηνική βόμβα, το Ιράν κατασκευάζει επιπλέον πυράβλους μεγάλου βεληνικούς ε, που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Έτσι μπορεί να φτάσει και σε μακρινές γωνιές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης. Πιστεύω ότι εκτός από τον έλεγχο της παραγωγής εμπλουτισμένου και μάλιστα υψηλό εμπλουτισμένου ουρανίου υπάρχει έλεγχος, ανάγκη να ελέγχεται και ο τρόπος ε, παραγωγής. Ε, η παραγωγή των ε, πυράβλων που είναι σε θέση να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Ο Χαμενεή δήλωσε ότι η θρησκεία απαγορεύει την παραγωγή όσο και τη χρήση πυρηνικών όπλων για ποιο λόγο κατασκευάζει πυράβλους που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Ενσίνκη που έλαβε χώρα το 1975, οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής έθεσαν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στη Σοβιετική Ένωση ως πρώτη προτεραιότητα ε, του κόσμου τότε. Αυτό προκάλεσε έκπληξη, αλλά ήταν και αποτελεσματικό. Δείχνει ότι η φωνή της ηθικής δεν είναι λιγότερο σημαντική από ε, τα διπλωματικά διαβήματα. Σήμερα η έκκληση αυτή θα πρέπει να απευθυνθεί προς το Ιράν. Μία σαφής φωνή θα πρέπει να ακουστεί κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ιρανικό καθεστώς. Μια σαφής φωνή θα πρέπει να ακουστεί κατά ενός καθεστώτος το οποίο απαγχωνίζει ανθρώπους χωρίς δίκη, που ρίχνει δημοσιογράφους στη φυλακή χωρίς δίκη που βάλει με πραγματικά πειρά κατά πολιτών, διαδηλωτών, χωρίς σεβασμό για τη ζωή τους. Μια σαφής φωνή θα πρέπει να ακουστεί κατά ενός καθεστώτος που ε, προχωρεί σε διακρίσεις κατά των γυναικών. Και αντί να μοιράζεται τα κέρδη από το πετρέλαιο με το λαό του, το καθεστώς αυτό το δαπανά ε, στη δημοκρατία, σε όπλα ε, που θέτει σε κίνδυνο λαούς σε όλο τον κόσμο. Το εμπλουτισμένο ουράνιο φτωχαίνει πεινασμένα παιδιά. Η φωνή της ηθικής θα εθαρρύνει τον Ιρανικό λαό στο δικό του αγώνα για ελευθερία, στη δική του πάλι κατά της φτώχειας. Πολύ σύντομα θα λάβουν χώρα εκλογές στο Ιράν. Δεν θα πρέπει να αφαιθούν οι αγιατολάδες να στρεβλώσουν και να νοθεύσουν τα αποτελέσματα. Να απογοητεύσουν και να κυρώσουν το δικαίωμα του λαού να κάνει τη δική του ελεύθερη επιλογή. Η δική σας φωνή, κυρίες και κύριοι, θα δείξει στον Ιρανικό λαό ότι η Φίλιος δεν τους έχει γυρίσει την πλάτη. Οι σημερινοί ηγέτες του Ιράν παραβιάζουν το χάρτη των ε, Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος καταδικάζει την παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων και την ε, εισβολή και επίθεση έναντι άλλων εθνών. Ωστόσο έχουν τη δυνατότητα ε, να καταχρώνται ε, αυτή τη διάταξη και μάλιστα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν υποστηρίζει την τρομοκρατία παντού στον κόσμο. Ο βασικός της αντιπρόσωπος, η Χεσπολάχ, εκτελεί τρομοκρατικές επιθέσεις και απειλεί τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής. Και αγαπητοί φίλοι, η ιστορική συμφωνία Σάιξ Πικό μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας γέννησε το σύγχρονο Λίβανο με σκοπό να γίνει μια χώρα πολυεθνική όπου μουσουλμάνοι, χριστιανοί και δρούζοι θα συμβιούν ειρηνικά. Σήμερα η Χεσμολάχ με την υποστήριξη του Ιράν καταστρέφει το Λίβανο. Η Χεσπολά είναι τρομοκρατική εργάνωση. Δεν είναι πολιτικό κίνημα. Συλλέγουν πυράβλους. Είναι πολεμοχαρείς. Κρύβουν πυράβλους σε ειρηνικά χωριά και πόλεις. Και πράττοντας έτσι γίνονται πολεμικοί στόχοι οι πόλεις και τα χωριά. Η Χεσπολά διαιρεί το Λίβανο πολιτικά, θρησκευτικά και εθνικά. Έχει μετατρέψει τη χώρα του κέντρου σε μια χώρα άγωνη και με ε, κέντρους κατεστραμμένους. Η είναι κράτος εν κράτη. Ε, είναι ένας ιδιωτικός στρατός στο περιθώριο του εθνικού στρατού στέλνει ε, στρατιώτες να υποστηρίξουν ε, τις φαγές ενός αιμοσταγού δικτάτορα στη Συρία χωρίς ε, έγκριση και άδεια της κυβέρνησης στην οποία συμμετέχουν. Πρόσφατα 20 τρομοκρατικές απόπειρες της Χεσπολάχ διεξήχθησαν παντού στον κόσμο. Ινδία, Ταϊλάνδη, Γεωργία, Νότια Αφρική, Ηνωμένε Πολιτείες, Αίγυπτο και Ελλάδα μεταξύ άλλων χωρών. Τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ταυτοποίησε ε, τους δράστες της τρομοκρατικής ενέργειας στο Μπουργκάς. Ε, και ήταν της Χεσμολάχ. Πέντε Ισραηλινοί τουρίστες και ένας Βούλγαρος πολίτης έχασαν τη ζωή τους. Πρόσφατα η Κύπρος συνέλαβε ένα τρομοκράτη της που σχεδίαζε τρομοκρατική απόπειρα. αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Απευθύνουμε έκκληση σε εσά. Να ονομάζετε την τρομοκρατία τρομοκρατία. Σώστε το Λίβανο από την τρομοκρατική τρέλα. Σώστε το λαό της Συρίας από τους αντιπροσώπους του Ιράν. Σώστε τους δικούς σας και τους δικούς μας πολίτες από τύχες πολλά. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να στιγματίσει τη Χεσμολάχ ως τρομοκρατική οργάνωση διότι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Σήμερα η τρομοκρατία απλώνει τα πλοκάμια της πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Πρόσφατα αποπειράθηκαν οι τρομοκράτες να ε, αναλάβουν την εξουσία στο Μαλί. Αν το είχαν επιτύχει θα είχαν σταματήσει τις εντυπωσιακές προσπάθειες ε, της Αφρικανικής Υπήρου να ανακάμψει από το παρελθόν της. Μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες για όλους εμάς είναι ε, το γεγονό ότι βλέπουμε θαραλέες προσπάθειες στο λαό της Αφρικής να δημιουργήσουν μια απο τις μεγαλυτερες ελπιδες για ολους εμας ειναι το γεγονος οτι βλεπουμε νέα που να βασίζεται στην επιστήμη όπως και στην Ευρώπη. Ο ελεύθερος κόσμος δεν μπορεί να παραμένει θεατής καθώς η τρομοκρατία βάζει χέρι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, του παλιού είτε του νέου, του κοντινού ή μακρινού. Δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές όταν ε, ο Σύρος Πρόεδρος ε, αφανίζει τον ίδιο του το λαό ε, και τα παιδιά. Πρόσφατα ο Άσαντ έκανε και πυρηνικό εργοστάσιο και ένα οπλοστάσιο χημικών όπλων ενώ το πυρηνικό εργοστάσιο κατεστράφει εγκαίρως, ε, το χημικό οπλοστάσιο παραμένει στα χέρια του τη στιγμή αυτή που μιλούμε. Είναι ε, τρομακτικός κίνδυνος για το λαό της Συρίας και για τη σύνολη περιοχή, ακόμα και για την Ευρώπη. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος για να μην πέσουν σε λάθος χέρια τα χημικά όπλα η καλύτερη λύση για να τερματιστεί η Συριακή τραγωδία θα μπορούσε να επιτευχθεί δίνοντα τη δυνατότητα στον Αραβικό Σύνδεσμο να παρέμβει, το οποίο μέλος του Αραβικού Σύνδεσμου είναι η Συρία. Ε, μία επέμβαση των δυτικών δυνάμεων ε, θα θεωρεί το ως ξένη ανάμιξη. Ο Αραβικός Σύνδεσμος μπορεί και θα έπρεπε να δημιουργήσει ε, μια προσωρινή κυβέρνηση στη Συρία για να σταματήσουν οι σφαγές, για να μην κατακαιρματιστεί η Συρία. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη θα έπρεπε να υποστηρίξουν ε, τον Αραβικό Σύνδεσμο για να δημιουργηθούν δυνάμεις Αράβων και Ανοκράνων. Αγαπητοί φίλοι, πριν από 18 χρόνια ήρθα στις Βρυξέλλες για να υπογράψω τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Χαίρομαι που η πραγματικότητα υπερεύει τις προσδοκίες μας. Είναι γεγονός ότι η Συμφωνία Σύνδεσης ε, έγινε εταιρική σχέση και εδώ και καιρό η εταιρική σχέση έχει γίνει φιλία. Σε αυτά τα γερά θεμέλια προτείνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ισραήλ να συνεργαστούν προς όφελος της σταθερότητας και της ευημερίας στη Μέση Ανατολή. και γενικότερα την ανάπτυξη και άλλων περιοχών του κόσμου. Το Ισραήλ περιγράφεται ως ένα έθνος νεοφανές ε, startup. Ελπίζω ε, και όλη η Μέση Ανατολή να γίνει τέτοια περιοχή ε, με υποστήρες υψηλή τεχνολογίας που θα μπορέσουν ε, να βοηθήσουν την περιοχή να ξεφύγει από τη φτώχεια. Είναι μικρό το Ισραήλ. Γι' αυτό προσπαθούμε το μέγεθός μας αυτό να το κάνουμε πλεονέκτημα ανακαλύψαμε ότι μικρές χώρες μπορούν να γίνουν μεγάλα πιλωτικά προγράμματα. Σήμερα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό πρότυπο που θα γεφυρώσει το χάσμα ε, ανάμεσα στους έχοντες και τους μη έχοντες. Το κοινωνικό χάσμα είναι μείζον πρόβλημα για όλους μας, φτωχούς και πλουσίους. Αναζητούμε νέους τρόπους να ξεπεράσουμε αυτό το χάσμα ε, με εκδημοκρατισμό της υγείας, της παιδείας, με εκδημοκρατισμό της τηλεπικοινωνίας και μείωση του κόστους ε, τροφής και στέγης. Είναι επιτακτική αυτή η ανάγκη για τη νέα γενιά. Ξέρω ότι είναι ωραίο να είσαι νέος, αλλά είναι και πανάκριβο προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρώπων. Να μπορεί ο καθής να έχει τη δυνατότητα να κάνει μια ελεύθερη επιλογή για τον τρόπο ζωής του. Και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε ε, διεισδύοντας στα μυστικά του εγκεφάλου μας. Ο εγκέφαλος είναι το πιο θαυμαστό εργαλείο στον κόσμο. Μας έχει δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τεχνητούς εγκεφάλους. Ωστόσο, απέχουμε ακόμα πόρο από την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ίδιου του εγκεφάλου. Ουσιαστικά, είμαστε οι ίδιοι. Είμαστε άγνωστοι, ξένοι για τον εαυτό μας. Ανακαλύπτοντας το μηχανισμό του εγκεφάλου μας, θα καταφέρουμε να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και με τον πλησίον μας. Χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια έχει καταστεί νέα προτεραιότητα και είναι ένα μείζον θέμα συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεών μας, των μη κυβερνητικών μας οργανώσεων και μεταξύ ημών ως ε, προσώπων και ετών. Ο παγκόσμιος κόσμος μας δεν έχει παγκόσμια διακυβέρνηση και μάλιστα ε, είναι σχεδόν ακυβέρνητος και δεν υπάρχει δυνατότητα να κυβερνηθεί. Θα πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική λύση. Εγώ πιστεύω ότι οι μελλοντικοί τρόποι διακυβέρνηση θα πρέπει να βασίζονται σε τρεις πυλώνες. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα εξακολουθούν να φέρουν ε, το βάρος της ε, αναπαραγωγής του κράτους έθνους. Ε, οι παγκόσμιες εταιρείες θα επενδύσουν στην έρευνα και την ανάπτυξη και το άτομο, ο καθένας ξεχωριστά, θα έχει τη δυνατότητα να κυβερνάει τον εαυτό του γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλός του. Σήμερα η επιστήμη λέει πολύ περισσότερα από την πολιτική είναι και παγκόσμια αλλά δεν γνωρίζει και σύνορα. Οι στρατοί δεν μπορούν να κατακτούν ε, τη γνώση και οι αστυνομίες δεν μπορούν να συλλαμβάνουν την επιστήμη. Εγώ πιστεύω στην επιστημονική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Παγκόσμιες επιστημονικές εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν για να αλλάξει ο κόσμος. Η παγκοσμιοποίηση έθεσε τέρμα στο ρατσισμό δεν μπορεί κανείς να είναι και παγκόσμιος και ρατσιστής. Η παγκοσμιοποίηση ε, δεν δυναμώνει το άτομο. Οι παγκόσμιες εταιρείε δεν επιβάλλουν τη βούληση τους σε λαούς. Το αντίθετο, σέβονται ε, τη βούληση των πελατών τους. Μπορούν να παράσχουν όμως ε, επιστημονική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη. Μπορούν να βοηθούν νέους να μορφώνονται σε πανεπιστήμια. Ε, μπορούν να δημιουργούν θέσεις εργασίας ανάλογες των προσόντων και των δεξιοτήτων τους. Αυτή είναι η καλύτερη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στη νέα γενιά μας και στον αραβικό κόσμο ε, για να μπορέσουν να απαντήσουν στις προκλήσεις της νέας εποχής και αυτή είναι η ελπίδα μας. Ε, πρότεινα ένα σχέδιο για μια κοινοπραξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ κυβερνήσεων, εθνικών κυβερνήσεων και παγκοσμίων εταιριών, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε ε, σε αυτές τις προκλήσεις με ένα νέο τρόπο. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζω ότι αυτό χρειάζεται την υποστήριξή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου να προσβλέπω στην κατανόησή σας όσο και τη βοήθειά σας. αν ενώσουμε τη γνώση της Ευρώπης με την εμπειρία του Ισραήλ, μπορούμε να υπερβούμε τις αυριανές προκλήσεις. Αντιμετωπίζοντας την έλλειψη μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης, μπορούμε να σφυριλατήσουμε στενότερη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και παγκοσμίων επιχειρήσεων. Αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους που απειλούν τις αξίες ε, ε, τις οποίες πρεσβεύουμε, θα καταπολεμήσουμε ε, χωρίς να αφιστούμε κόπον ε, τη τρομοκρατία όπου και αν βρίζεται. Πρόεδρε Σούλτς, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Ο Ζάμονε, ο πατέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε πει κάποτε «Φιλόδοξοι είναι όλοι. Το θέμα είναι αν είσαι φιλόδοξος να είσαι ή αν είσαι φιλόδοξος να πράτης. Έχει έρθει η αν εισαι φιλοδοξος να πραττεις εχει ερθει η ωρα των πράξεων ας μην λησμονούμε ότι είμαστε τόσο σπουδαίοι όσο ο σκοπός τον οποίο υπηρετούμε. Βεβαίως είναι τρομακτικές οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά ποιος είναι καλύτερα σε θέση να αντιμετωπίσει το φαινομενικά αδύνατο από δύο θαύματα, τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ για να αντιμετωπίσουμε και να υλοποιήσουμε τις διδαχές της ε, κληρονομιάς μας. Με τα λόγια των ε, προκατόχων μου και των προγόνων μου, ας διορθώσουμε τον κόσμο. Τικούν ολάμ, λέγεται στα εβραϊκά αυτό. Με τα λόγια του Ζαμονέ, ας πούμε, ας πράξουμε επιτέλους. Ας συνεργαστούμε για μια καλύτερη Μέση Ανατολή με μια Ευρώπη θαραλέα και τολμηρή. Ας υλοποιήσουμε τις αξίες των λαών μας. Ειρήνη, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα. Να μην ε, λιγοψυχήσουμε σε κανένα εμπόδιο, να τολμήσουμε το νέο. Θα πρέπει να είμαστε υπηρέτες του μέλλοντος αντί αφέντες του παρελθόντος. Αγαπητοί φίλοι, βλέποντας το μέλλον της φιλίας μας, του Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι γεμάτος ελπίδης και αποφασιστικότητα. Χέρι με χέρι θα χτίσουμε ένα καλύτερο και πιο φωτεινό αύριο για τις αυριανές γενναίες. Σας ευχαριστώ πολύ και σαλόμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι για την τιμή που αποτίσατε στον Πρόεδρο Πέρες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα λόγια σας. Νομίζω ότι η έκκληση που απευθύνατε σε μας θα γίνει εισακουστή. μεταξύ του λαού του Ισραήλ και του λαού των ευρωπαϊκών χωρών υπάρχουν οι δεσμοί που αναφέρατε και ο σεβασμός για το άτομο και την απαράγραπτη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτό ισχύει και για την Ευρώπη και για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη και για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ.